Uh, well, good morning everybody. Um, welcome to um, our... Um, Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, τη δημόσια συνεδρίασή μας. Με την ε, μετάδοση μας του διαδικτύου, με δύο θέματα, επαγγελματικές δεξιότητες και ενιαία αγορά. Με τον κύριο Για να μην καθυστερούμε λοιπόν. Παρακαλώ τον εισηγητή για την πολύ σημαντική αυτή πρόταση για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τις επαγγελματικές ε, για τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες. Και έχουμε και θέματα βέβαια να δούμε με τις συμβαστικές τροπολογίες, πότε θα τα κτλ. από την Επιτροπή. Δεν βλέπω τον κύριο Τίτσερ εδώ. Αλλά κάποιος από τους συναδέλφους τους θέλησουν να συμμετάσχουν. Οι σκιώδεις ηγητές μας είναι παρόντες. Και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την κυρία Βερνιό να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις και στη συνέχεια στους σκιώδεις ηγητές. Περνάτε, έχεις το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Il y a trois semaines, nous avons... ε, ξεκινήσαμε λοιπόν με τους συναδέλφους σκιώδης εισηγητές να εκμεταλλευόμαστε την παράταση που είχαμε ζητήσει. Θα ήθελα δε ιδιαίτερω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα των σκιωδών εισηγητών και φυσικά και τους ε, βοηθούς τους, όλο το προσωπικό το οποίο συνεργάστηκε μαζί μας, γιατί δουλέψαμε σε πολύ επικοδομητικό ε, ε, κλίμα και αυτό είναι πολύ καλά. Ε, κάναμε λοιπόν ε, τακτικές ε, προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τρόπο ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στην συνάντηση των σκιωδών. Θα είμαι μάλλον σύντομη σήμερα γιατί νομίζω ότι, ήδη, ότι κάποιοι βουλευτές δεν είχαν εκτός των σκιωδών τη δυνατότητα να μιλήσουν όσο ήθελαν. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ μονάχα με μερικά σημεία στα οποία πλησιάζουμε. Ε, σε συμβιβασμό. Όσον αφορά την μερική πρόσβαση, ε, θέλουμε ε, να έχουμε πολύ καλή πλαισίωση αυτού του ζητήματος και το κράτος υποδοχής να μπορεί να αποφασίσει βάσει κανόνων που διέπονται από τους κανόνες του εθνικού συμφέροντος και να πούμε οπωσδήποτε ότι ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μονάχα μετά από άρνηση της πλήρους αναγνώρισης. Όσον αφορά την επαγγελματική κάρτα, όλοι θέλουμε να τροποποιήσουμε τις προθεσμίες έτσι ώστε ε, να ε, δοθεί περισσότερος ο χρόνος βέβαια στις διοικητικές αρχές, αλλά αυτός ο χρόνος να μην είναι υπερβολικός χρόνος αναμονής για τους επαγγελματίες και ε, βεβαίως να μην ξεπερνιούνται αυτές οι χρονικές προθεσμίες. Επίσης, οδηγούμαστε σε ε, συμφωνία όσον αφορά τον καθορισμό του τι καλύπτουν τα στάζ, αυτές οι ταχύριθμες εκπαιδεύσεις στα πλαίσια της οδηγίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολυάριθμους νέους που ακολουθούν τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις στάζ. Ο μηχανισμός ε, προειδοποίησης ε, είναι κάτι σημαντικό. Μας ε, ενδιαφέρει πολύ και προσπαθούμε να τηρήσουμε όλες τις εθνικές συνήθειες. Είτε αφορούν τον περιορισμό, είτε την απαγόρευση πρόσκαιρη ή μόνιμη άσκησης του επαγγέλματος. Όσον αφορά το ζήτημα των γλωσσικών εξετάσεων, των δοκιμασιών αυτών. Βεβαίως μελετήσαμε το θέμα του κόστους και εδώ ακόμα το συζητούμε βεβαίως, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εξέβρεση συμφωνίας. Συζητούμε, λέω, για τις ε, ε, που παρουσιάζουν οι χώρες με ε, περισσότερες από μία γλώσσα, ας πούμε στο Βέλγιο, φλαμανδικά και γαλλικά, ε, στην Ισπανία, ε, ε, ισπανικά και καταλανικά κτλ. Νομίζω ότι εδώ έχουμε περιθώριο να βρούμε σημεία ισορροπίας σημειώστε ότι δεν είναι τα πιο ε, σημαντικά ή διχαστικά στοιχεία γιατί ε, εμείς τώρα θα ασχοληθούμε και με άλλες οριζόντιες υποθέσεις, άλλα οριζόντια ζητήματα και βεβαίως θα δούμε ε, και τομεακά ζητήματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένα επαγγέλματα γιατί έχουμε κάποιες δυσκολίες όσον αφορά κάποια επαγγέλματα παρά τα αυτά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Να σας πω λοιπόν ότι προσωπικά ε, σήμερα δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα των νοσηλευτριών Βεβαίω εσεί μπορείτε να το αναφέρετε αν θέλετε, δεν μπορώ να σα το απαγορεύσω. Πιστεύω ότι το ζήτημα των ε, νοσηλευτών θα πρέπει, ε, να, ε, θα πρέπει σε αυτό το ζήτημα να ησυχάσουν λίγο τα πνεύματα. και η Κυπριακή Προεδρία και η μελλοντική Ιρλανδική Προεδρία, την οποία συνάντησα και η οποία θεωρεί πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Συζητούν λοιπόν οι Προεδρίες, η σημερινή και η μελλοντική, το θέμα στο Συμβούλιο. Βρίσκομαι σε τακτική επαφή μαζί τους αλλά και με την Εκτελεστική Επιτροπή. Γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι σημαντικό στο μέτρο ε, που η Κομισιόν και το Συμβούλιο είναι οι εταίροι μας ε, στον καθορισμό μιας, ε, ενός καταλόγου ικανοτήτων που ακόμα δεν μας ικανοποιεί. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε αφήσουμε λίγο το ζήτημα αυτό στην άκρη, ε, να κατευναστούν λίγο τα πνεύματα και να ασχοληθούμε εντωμεταξύ με τα άλλα ζητήματα, τα οποία είναι εξίσου φλέγοντα. Τούτη τη στιγμή και λαμβάνοντα υπόψη την παρούσα κατάσταση, γιατί βεβαίω έχουμε ε, την ε, Κομισιόν η οποία έχει καθορίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο κείμενό τη, ξέρουμε ε, πώ έχουν τα πράγματα, θέλουμε μια εναρμόνιση προ τα πάνω. Παρόλα αυτά υπάρχουν χώρε οι οποίε αντιμετωπίζουν δυσκολίε όπω ξέρετε και οι οποίε μα θέτουν και εμά κάποια προσκόμματα και επομένω ναι, μεν θέλουμε να βρούμε συμφωνίε και συμβιβασμού, αλλά ικανοποιητικού συμβιβασμού Κατά την άποψή μου, αυτό που πρέπει να ε, μας απασχολεί είναι οι ίδιοι οι επαγγελματίε, οι νοσηλεύτριε, είναι ένας τομέας με μεγάλο βαθμό κινητικότητας. Ε, γιατί ας πούμε ε, το ποσοστό κινητικότητας των συμβολεογράφων είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τους συμβολεογράφους, ε, καθόλου μάλιστα. Αλλά στο θέμα, στο επάγγελμα των νοσηλευτών, η κινητικότητα είναι εξαιρετικά μεγάλη και δεν θέλουμε να πάρουμε καμία απόφαση η οποία θα ενισχύσει την ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν ε, αυτοί οι εργαζόμενοι. Αυτά λοιπόν και ευελπιστώ ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε ένα κείμενο το οποίο μπορεί θα μπορεί μάλλον να διασφαλίσει την επαγγελματική κινητικότητα χωρίς όμως να ζημιώνει καθόλου η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι πολίτες και οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Μπερναντέτ για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι σκιώδεις εισηγητές. We still have to get to grips with. Um, ε, Merci, Monsieur le Président. Κυρία Λεγκρίπ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βερνιό και να πω ότι συμμερίζομαι τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε το, ε, την ατμόσφαιρα των ε, συναντήσεων μεταξύ εισηγητών, σκιωδών εισηγητών κτλ. Ε, ήταν πολύ επικοδομητικό αλλά και φιλικό και αυτό ισχύει σε κάθε μία από τις συναντήσεις μας. Για την ώρα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο έχουν προχωρήσει οι εργασίες, αλλά και με την παρουσίαση που μόλις έκανε η εισηγήτριά μας. Ε, υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί οι οποίοι ε, είτε είναι έτοιμοι να αποδώσουν, είτε έχουν, βρίσκονται σε πολύ προωθημένο βαθμό προετοιμασίας. Ε, είναι γεγονός ότι έχουμε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου για να ε, συνεχίσουμε την εργασία ε, και την εργασία τη δική μου στην εκπροσώπηση της ομάδας μου για να ε, υποβάλουμε την εργασία μας, την έκβαση των εργασιών μας στην Επιτροπή. ναι, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα και όσον αφορά την απαραίτητη ευελιξία έτσι ώστε να βρούμε τον τρόπο για να βάλουμε το σωστό κέρσορα στο σωστό σημείο για να βρούμε το, την, το σωστό χρονικό περιθώριο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία νομίζω είμαστε έτοιμοι να τα λύσουμε. Επαναλαμβάνω ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει και ε, εργαλείο, ε, όπλο ε, διαπραγματευτικό στις διαπραγματεύσεις μας. Γιατί αυτό που θέλει το Κοινοβούλιο είναι να υποχρεώσει τις χώρες μέλη να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μεταξύ μας θα μπορέσουμε να έχουμε φτάσει σε μια καλή συμφωνία, σε έναν καλό συμβιβασμό ε, ε, ναι, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια περιθώρια ανέρεσης σε περίπτωση ε, αιτήματος περαιτέρω εγγράφων ή δικαιολογητικών κτλ. Το ζήτημα των προσόντων επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί η αναγνώριση των προσόντων δεν μπορεί να σημαίνει αυτόματα και αναγνώριση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος. Και βεβαίως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι και οι αρμόδιες αρχές ε, μέσα σε μια εβδομάδα θα μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Όσον αφορά τώρα ε, την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα σε ευρύτερο πλαίσιο, νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε κυρίως το ζήτημα των κέντρων αρρωγής και των σημείων επαφής. Υπάρχει η τροπολογία 230 του συναδέλφου Αρίας και η 229 της υποφαινομένης όσον αφορά αυτά τα κέντρα αρρωγής, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, εμπλακούν ε, στο παρασκευαστικό σχέδιο μαζί με τα σημεία επαφής. Ε, και θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα και τις αρμοδιότητες τις κατάλληλες για να δώσουν αυτήν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Προσώπων. Ε, όσον αφορά τα υπόλοιπα, την αναπερίπτωση ε, μελέτη κτλ. Έχω υποβάλει τροπολογίες και νομίζω ότι μπορώ να είμαι ικανοποιημένη με την εργασία που έχει μέχρι τούδε επιδευθεί, καθώς επίσης και με την εισαγωγή της έννοιας του κοινού συμφέροντος, διεθνή ωφελία, έννοια την οποία εγώ είχα ζητήσει ε, να ε, αναφερθεί. Voyons un peu plus euh, précis, un peu plus... Ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ε, συγκεκριμένοι όσον αφορά ε, τον ορισμό του στάζ, τι είναι αυτή η εκπαίδευση στάζ. Νομίζω ότι το να, ακολουθήσουμε τα όσα αναφέρονται στην οδηγία για τα στάζ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και η αντιμετώπιση ήταν ομόφωνη στην ομάδα. Θα επιθυμούσα Πάντως, έστω και αν ήταν λίγο υπερβολικά συγκεκριμένες οι τροπολογίες που έχω υποβάλει, θα επιθυμούσα παρόλα αυτά να καταφέρουμε να καθορίσουμε ε, τις μεγάλες γραμμές ενός πλαισίου ποιότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους νέους μας, ε, για τους νέους πολίτες, τη νέα γενιά. Δηλαδή, ίσως ένα κανονικό άρθρο και όχι μια απλή αιτιολογική σκέψη να προσπαθήσει να αποσαφηνίσει τα ζητήματα αυτά. Ε, γλωσσικές ικανότητες. Νομίζω ότι θα επιτύχουμε συμφωνία. Ήταν ένα ζήτημα επί των οποίων ε, πολλά μέλη της πολιτικής μου ομάδας ε, είχαν εκφράσει ανησυχία και προβληματισμό. Για την ώρα νομίζω ότι σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι μία Μία μονάχα γλώσσα, ε, γνώση γλώσσας χρειάζεται για τις χώρες, ε, ε, για, την πρόσβαση στα επαγγέλματα στις χώρες οι οποίες έχουν ε, περισσότερες από μία γλώσσες. Η αναφορά στο άρθρο 53.2 ε, νομίζω ότι ε, όσον αφορά τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες νομίζω ότι μπορεί να είναι ολιστηρός ο δρόμος αυτός και μπορεί να οξύνει κάποια πνεύματα ήδη οξυμένα. Όσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες τις οποίες ανέφερε η κυρία Βερνιό, έστω και αν δεν θέλει να διονγκωθεί και να ξανασυζητηθεί και να ξανασυζητηθεί γιατί όντως χρειάζεται κάποια ηρεμία πνεύματα τόσο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις ε, ε, εργασίες μας. Το, το, επάγγελμα των συμβολιογράφων και των νοσηλευτών νοσηλευτηριών. Ε, πρέπει να πω για τους μεν συμβολιογράφους ότι δεν έχουμε απλώς παροχή υπηρεσιών, δεν είναι απλή παροχή υπηρεσιών. Νομίζω ότι έχουμε εδώ εκπροσώπους της, των δημοσίων αρχών ε, στο, στην περίπτωση των συμβολιογράφων. Επομένω, θα πρέπει ιδιαίτερω να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε αυτού του επαγγέλματο. Υπενθυμίζω δε ότι ο αριθμό των κρατών στι ευρωπαϊκέ ε, χώρε δεν γνωρίζουν του που δεν, δεν έχουν δηλαδή του συμβολιογράφου αστικού δικαίου ε, είναι μειοψηφία. Είναι πολύ λίγε. Ακόμα και η Κροατία που είναι το καινούριο μέλο λειτουργεί με αυτό το σύστημα του συμβολιογράφου αστικού δικαίου. Ε, τώρα, όσον αφορά ε, όσον αφορά τα όσα αναφέρει η συγγήτρια στο προσχέδιο, ε, δεν είμαι απολύτως πεπισμένη. Βεβαίως ακούω προσεκτικά, ακούω και τους συναδέλφους, βλέπω τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Μερικές μάλιστα έχουν υποβληθεί από έγκριτα μέλη της ομάδας μου ε, ε, πολλοί μεταξύ αυτών έχουν επιλέξει ε, μια διαφορετική γραμμή, δηλαδή θέλουν διαχωρισμό ανάμεσα στην ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος. Εν πάση περιπτώσει θα τα ξαναδούμε αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση stand still. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Θα δούμε ποια θα είναι η λύση. Θα βρούμε μια λογική λύση για μια ακόμα φορά. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην, ε, ε, να, μην δείξουμε έλλειψη σεβασμού προς ε, παραδόσεις ετών. Όσον αφορά νοσηλευτές, νοσηλευτριές, άλλο ευαίσθητο θέμα, υπενθυμίζω ότι η ομάδα ΕΛΚΕ έχει υποβάλει τροπολογία η οποία κατά την άποψή μου είναι και συμφιλιωτική και συνθετική και επικοδομητική, βάσει του άρθρου 31, τροπολογία μέσα στην οποία η ομάδα μου ε, αναφέρεται στους ε, δύο πυλώνες, αυτό το διτό σύστημα, dual system. Ε, γνωρίζω βεβαίως ότι η παρούσα εκδοχή αυτής της συμβαστικής τροπολογίας της ομάδας μου δεν έχει πείσει ακόμα την εισηγήτρια, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί βάση συζήτησης. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εργασία σε βάθος έτσι ώστε να δούμε τον κατάλογο κυρίως των προσόντων. Υπάρχει και η Επιτροπή ΕΝΒΗ Περιβάλλοντος η οποία ε, πρέπει να εκπονήσει γνωμοδότηση. Γνωρίζω ότι κατά μεγάλη πλειοψηφία έχει συμφωνήσει ε, υπέρ των 10 ετών κατάρτισης για τους νοσηλευτές. Νομίζω ότι και εδώ μπορούμε να βρούμε την χρυσή τομή. και, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε ε, να μην μπερδευτούμε με πολλά πράγματα Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, λέω, έτσι ώστε να μην θέσουμε εν αμφιβόλο την νομιμότητα των συστημάτων κατάρτισης που έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι σωστά, ε, που σε πολλές χώρες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, αν όχι εδώ και ε, εκατονταετίες, εδώ και αιώνες και που έχουν δημιουργήσει γενιές και γενιές ανθρώπων πολύ ικανών. Ε, και όλα αυτά να τα κάνουμε στο όνομα της ε, ε, ομοιογενοποίησης, της εναρμόνισης των ικανοτήτων και τα λοιπά. Και το ζήτημα του vocational training, νομίζω ότι, που έχει προσυπογραφεί από πάνω από 10 βουλευτές, νομίζω ότι επίσης πρέπει να μας απασχολήσει και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά και χαίρομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμο η απόψεις σας και η θέση σας. Ο κύριος Μπουζόη. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Βερνιό και του ε, λοιπού και ηγητές, ε, την κυρία Ντεκλίπ ε, και όλου του άλλου και ηγητές με του οποίου συνεργαστήκαμε. Είχαμε κάποιε συνεδριάσει των νησμού. Όπως είπε και η κυρία Βερνιά, το προσωπικό μα παραμένει σε επαφή ακόμη. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδο των εργασιών στο θέμα αυτό και θα είμαι σύντομο, καθώ ήδη έχω τοποθετηθεί αρκετέ φορέ. για τα θέματα είτε των, ε, του ελέγχου των γλωσσικών γλώσσεων, των γλωσσικών γνώσεων, είτε των συμβολιογράφων. Θα ήθελα να αφαιρθώ ωστόσο στο 43β την τροπολογία που έχω, καταθέσει και τα συζητήσει με τις ε, αρχές της Ρουμανίας διαπιστώνουμε ότι δεν χρειάζεται πλέον η κατάργηση του εν λόγω άρθρου. Αφορά τις ΜΕΕΣ, όχι τις νοσηλεύτερες αλλά τις ΜΕΕΣ οι οποίες είναι περιορισμένα στον αριθμό, έχουν παλαι... απεπαλαιωμένα διπλώματα γιατί το 1982 βγήκαν οι τελευταίες από τη σχετική σχολή. Επομένω, τα διπλώματά του είναι παλαιά. Άρα πλησιάζουν λίγο πολύ οι διπλωματούχοι ε, με ε, την ε, ηλικία της ταξιοδότησης, εξού και δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη για τα θέματα της κατάρτισης, όπως στο θέμα των νοσηλευτριών. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο και αποσύρω την τροπολογία μου, πλην όμω εμένω στην ε, τροπολογία για κατάργηση 33β, του 33β, γιατί η κατάσταση που αφορά τις νοσηλεύτρες είναι ριζικά διαφορετική. Το έχω ήδη εκθέσει και στην Επιτροπή. Έχω καταθέσει το σχετικό έγγραφο που εξηγεί λεπτομερώς την κατάσταση των νοσηλευτριών στην ε, Ρουμανία. Ελπίζω ότι θα ήταν χρήσιμο για να σχηματίσετε μια εικόνα της κατάστασης. Θα ήθελα όμως να περάσω και σε κάποια σχόλια για το θέμα της αυτόματης αναγνώρισης για τα επαγγέλματα υγείας. Γιατί όπως είπε και η κυρία Βεγνιώ σε μια προηγούμενη συζήτηση, Έχουμε και άλλες τροπολογίες που αφορούν το 76 του σχεδίου κανονισμού που στόχο έχει να περιορίσει το καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης σε περίπτωση όπου ο επαγγελματίας δεν έχει ασκήσει για συγκεκριμένο αριθμό ετών την επαγγελματική του δραστηριότητα. Εξακολουθώ να πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι καλή ιδέα. Δεν πρόκειται για πρόοδο αλλά για οπισθοδρόμηση και θα επιδεινώσει την, ε, το γραφειοκρατικό βάρο φόρτο για την άσκηση ενό επαγγέλματο. Ένα ιατρό, για παράδειγμα, που έχει εξασκήσει το επάγγελμα επί 15 χρόνια, δεν χάνει τις, τις ικανότητες του επειδή μετά ενδεχομένως σταμάτησε να δουλεύει για 13 χρόνια ή λιγότερο. Ίσως για κάποιους άλλους λόγους, επαγγελματικούς, οικογενειακούς, προσωπικούς, δεν θα μπόρεσε να δουλέψει και θα πρέπει γι' αυτό να τον τιμωρήσουμε αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε ένα ορατό σε ένα καθαρό πλαίσιο, να δεχόμαστε βέβαια και να προωθούμε τη συνεχή διαρκή κατάρτιση και πάνω απ' όλα πρέπει αυτή η διαρκή κατάρτιση να την χάνει αναγνώριση αμοιβέ μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαιτέρω δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί συμβασμό για το θέμα των νοσηλευτριών. Συμφωνώ με την κυρία Βερνιό προσωπικώ και πιστεύω ότι ο στόχο μα θα πρέπει να είναι να συγκλίνουμε προς ένα κοινό ε, καθεστώς προς όφελος βεβαίως των επαγγελματιών χωρίς να πιστεύω ότι ένα διπλό, ένα διτό σύστημα θα μπορούσε να είναι χρήσιμο μπορώ να δεχθώ να το συζητήσω γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η ε, Γερμανίδες νοσηλεύτες, σε παραδείγματι, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποιες τέτοιες δυσκολίες. Ε, ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Συγήτρια και όλους τους συναδέλφους για τη διάθεση για συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω τώρα. Θα πάω στη Ρουμανία γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε εκλογές. Παραμένω όμως ψυχείτε και όχι σώματι στο πλευρό σας για την συνεργασία αυτή. Thank you very much. I know that... Uh, ε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι όλοι οι σκιώδεις συζητητές δουλεύουν πολύ σκληρά μαζί με την κυρία Βερνιό. Ευχαριστούμε πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας ε, για όλα αυτά που μας είπατε. Η κυρία Τούρνεν. Και εμείς ε, είμαστε ικανοποιημένοι με την συνολική εξέλιξη Εμείς ως πράσινοι έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση για να έχουμε καλύτερη κινητικότητα, αλλά να μην συμβιβαζόμαστε για ζητήματα όπως η υγιεινή, η ασφάλεια, η ε, καταλληλότητα των επαγγελματικών προσόντων και το γενικό όφελος βέβαια ε, κάτι το οποίο μπορεί να είναι πιο σημαντικό σε μερικές περιπτώσεις ε, από το να επιτρέψει κανείς την κινητικότητα. Οπότε πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία εκεί και πιστεύω ότι πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι κάνουμε ένα προσεκτικό βήμα. Νομίζω ότι ως κοιόδες εισηγητές ε, συγκλίνουμε σιγά σιγά και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είναι κάτι το οποίο έχει ε, αναγνωριστεί από το δικαστήριο. Πρέπει και εμείς να το αντιμετωπίσουμε, ε, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, ειδικότερα ως προς τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Όσον αφορά τώρα τις ε, προθεσμίες και την σιωπηλή αδειοδότηση, ε, πρέπει να πω ότι προσπάθησα να εξετάσω τι είναι το πιο κατάλληλο και τι είναι δύσκολο να τι θα πει δηλαδή κατάλληλη προθεσμία για να ζητήσουμε από τις αρχές να απαντήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από δύο μήνες ε, σε δύο εβδομάδες πάμε ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι τεράστιο βήμα. Οι αρχές, οι εθνικές λένε ότι θέλουμε βέβαια να επισπεύσουμε τη διαδικασία, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα μειονέκτημα γιατί δεν μπορούμε τελικά να τηρήσουμε τις προθεσμίες. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι ρεαλιστικό και πρέπει να δούμε ε, και τι πόρους έχουμε. Νομίζω ότι δεν είναι λοιπόν ιδεολογικό το ζήτημα, είναι κυρίως πρακτικό το ζήτημα του τι ακριβώς είναι η κατάλληλη προθεσμία. Εγώ είμαι ανοιχτή ε, ως προς αυτό. Τώρα έχουμε τις τρεις ε, εβδομάδες, το Συμβούλιο λέει τέσσερις εβδομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τους ανθρώπους ε, που όντως τα εκτελούν και δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση ε, στην οποία οι προθεσμίες θα είναι πάρα πολύ στενές. Όσον αφορά τώρα τις μαθητείες, την εκμάθηση, τα στάζ, ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερως που έχει συμπεριληφθεί αυτή η πρόταση, την οποία υποβάλαμε ως τροπολογία. Είπαμε ότι όταν είναι υποχρεωτικό τμήμα της κατάρτισης με σκοπό την πρόσβαση ή τη δυνατότητα ύπαρξης δικαιώματα ρύθμισης ενός επαγγέλματος, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να έχει να κάνει με την ε, επαγγελματική σου κατάρτιση, δεν πρέπει να είναι μια γενική φύσεως μαθητεία που δεν έχει καμία σχέση, γιατί βλέπουμε μια τεράστια έκρηξη αυτού του συστήματος που σημαίνει ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται από το επάγγελμά τους. Θέλουμε λοιπόν να είναι άμεση σχέση με το επάγγελμα και Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτό συμπεριλήφθηκε. Ε, όσον αφορά τώρα το πλαίσιο ποιότητας για τη μαθητή αυτή, Υπάρχει μια δεύτερη φάση διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου, την οποία δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μαθητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, αξιοπρεπή μαθητεία και ε, συνθήκε εργασία, αλλά αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε και σε άλλα σημεία. γιατί σε αυτή την οδηγία δεν ασχολούμαστε με τι συνθήκε εργασία, αλλά με το, το δικαίωμα άσκηση ενό επαγγέλματο ε, και την αναγνώριση ενό επαγγέλματο, τέλο πάντων των επαγγελματικών προσώπων, προσόντων συμφωνώ με την πρόθεση 100% και είμαι ανοιχτή σε κάθε πρόταση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η σωστή, το σωστό κείμενο να το ε, συμπεριλάβουμε. Επίσης ε, πρέπει να υπερβούμε και αυτό το δεύτερο στάδιο των διαβουλεύσεων γιατί πρέπει να δώσουμε και το δικαίωμα στους κοινωνικούς εταίρους να ε, εισακουστούν. Είναι δύσκολο θέμα, έχουν ένα δικαίωμα λοιπόν εκείνοι πρώτοι να διαπραγματευθούν, και είναι και ζήτημα επικουρικότητας. Ε, δεν υπάρχει μεγάλη αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρξει κανονισμός για τις συνθήκες εργασίας. Πρέπει να το πούμε και αυτό αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να απομακρύνουμε το δικαίωμα από τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευτούν εκείνοι πρώτοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό και για τους νοσηλευτές. Τέλος, νομίζω Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εδώ η συνάδελφος ε, θεωρεί και εκείνη ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε ένα καλό σύστημα. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε το γερμανικό σύστημα. Ο στόχος μας δεν είναι αυτός, αλλά να βρούμε μία λύση στα κενά που υπάρχουν, στο χάσμα που υπάρχει. Πρέπει κάπως να τα γεφυρώσουμε αυτά τα χάσματα μεταξύ ε, των 10 ετών και των 12 ετών ε, νοσηλευτών. Κάποιου είδους ε, μέτρα αντισταθμιστικά πρέπει να βρούμε. Κάποιο τρόπο τέλος πάντων να γεφυρώσουμε το χάσμα. Α, και για το μηχανισμό ειδοποίηση. Και εμείς είμαστε, και γι' αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, τη στιγμή που υπάρχει ένας περιορισμός ε, ή ε, ε, αν κάποιος ας πούμε δεν μπορεί πια να ασκήσει το επάγγελμα σε μια χώρα πρέπει να ενημερώνεται και η άλλη χώρα, ε, να υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία σε ένα σύστημα για να μπορέσει να το, ξέρει και, να το ξέρουν και οι άλλες χώρες. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάντελ είναι εδώ και η κυρία Μακλάρκιν είναι εδώ. Πρώτα η κυρία Μακλάρκιν, θα έλεγα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ 57 τροπολογίες υπέβαλα σε αυτή την έκθεση, οι οποίες ε, συζητήθηκαν ε, και στις προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων, αλλά θα ήθελα να επανεπισημάνω ορισμένα από τα βασικά σημεία που με απασχολούν. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις βάσει των συμβιβαστικών τροπολογιών για το γλωσσικό έλεγχο. Είμαστε σχετικώς ικανοποιημένοι με την κατεύθυνση που πήρε ο συμβιβασμός, αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε στο ότι θα έπρεπε να είναι δωρεάν ε, για όλους τους ετούντες. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει κάποια ευελιξία για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και το κόστος που συνεπάγεται αυτός ο γλωσσικός έλεγχος στα κράτη-μέλη. Ε, υπέβαλα μια τροπολογία που ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εποπτεύουν ε, επίσης, όχι μόνο δηλαδή να διενεργούν εκείνες τους ελέγχους ε, και θα ήθελα να μου πει η συγγήτρια κατά πόσο αυτό καλύπτεται παρκώς από τη συμβαστική τροπολογία τη σχετική και ποια είναι η άποψη της εισηγήτριας για την αξιολόγηση από πλευράς των αρμοδίων, ε, των αρμοδίων αρχών ε, πριν από την άσκηση του επαγγέλματος, ε, αλλά μετά την απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων. Συμφωνώ με την κυρία Τουρούνεν απολύτως ότι πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναστολής και αν θέλουμε να πιέσουμε σε σχέση ε, με ε, την ασφάλεια και τη υγεία. Νομίζω ότι οι προθεσμίες είναι πολύ ε, σημαντικές, αλλά υπάρχει και το σύστημα IMI, το οποίο πρέπει να συμμετέχει τη στιγμή της αναστολής να υπάρχει και μια ειδοποίηση αν έχουν χρησιμοποιηθεί παραποιημένα έγγραφα. Και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την επαγγελματική κάρτα, θα ήθελα να, με να ρωτήσω την ε, εισηγήτρια αν μπορεί να λάβει υπόψη την τροπολογία μου 271 για την ε, πιλωτική ε, προσπάθεια και την ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας. Η... Ε, Επιτροπή μίλησε για μια επαγγελματική, για μια εθελοντική, προαιρετική επαγγελματική κάρτα συμφωνούμε με την ιδέα, αλλά θα ήθελα αυτή η μερική πρόσβαση, ε, να μου πει η συγγήτρια αν θα μπορούσε να ισχύει όχι αναπερίπτωση, αλλά ένα επάγγελμα. Γιατί υπάρχει, ειδικά για όσους ασχολούνται με την ιατρική ε, φροντίδα, υπάρχει μια εξαίρεση στη συμβιβαστική τροπολογία και αυτό ίσως θα έπρεπε να ενισχυθεί για να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους στο πλαίσιο της, ε, των επαγγελμάτων της ιατρικής φροντίδας. Η βασική προτεραιότητα είναι η αναγνώριση ορισμένων ε, ε, επαγγελμάτων που δυσανάλογα μπλοκάρουν την πρόσβαση στα διάφορα κράτη-μέλη και πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά τα θέματα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κινητικότητα και την ανάπτυξη να επισπεύσουμε τις διαδικασίες στα κράτη-μέλη, ε, να μην μπλοκάρουν την πρόσβαση για λόγους ε, διαμονής ή ηθαγένειας και θα πρέπει να υπάρχει και ένας λόγος αν συμβαίνει αυτό που έχει να κάνει με το ε, δημόσιο συμφέρον τουλάχιστον. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, πιστεύουμε ότι μπορούμε να το ε, ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατόν και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να εστιαστούμε στο τι ακριβώς αφορά αυτό το νομοθέτημα, ε, την αναγνώριση και να επιτρέπεται η κινητικότητα των ε, επαγγελματιών. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι η πρόθεση αυτής της διαδικασίας για να μπορούμε ως, όσο το δυνατόν να ευθυγραμμιστούμε με τις απόψεις των ε, συνομιλητών. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Με ενθαρρύνει ο τρόπος με τον οποίο ε, συνεργάζονται οι, οι σκιώδεις και έτσι διευκολύνουν και επιταχύνουν ε, τους ρυθμούς των εργασιών. Τώρα βλέπω το κύριο Χέντελ είναι εδώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω αναλάβει στην πορεία του έργου τα καθήκοντα του κύριου Γκούστευσον. Γι' αυτό στο συγγνώμη αν τυχόν δεν είμαι σε θέση πάντοτε να είμαι 100% ενήμερος. Αλλά πρέπει να πω ότι γνωρίζω το θέμα αρκετά καλά. Πάντως, ζητώ συγγνώμη αν τυχόν τροπολογίες που έχω καταθέσει δεν είναι ακριβώς ε, εύστοχες ή ποιοτικέ. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα των ε, ε, νοσηλευτριών. Για το θέμα καταρχάς της μερικής πρόσβασης δεν είναι για μένα νοητό όσον αφορά τα ιατρικά επαγγέλματα εκτός και αν συμπληρωθεί η κατάρτιση με μια ειδική κατάρτιση η οποία θα συμπλήρωνε αυτή μερική τις μερικές δεξιότητες, τη μερική κατάρτιση. Ε, και εδώ έρχεται το θέμα της ασφάλειας των ασθενών στα επαγγέλματα της υγείας. Ιδιαίτερα σημασία πρέπει να αποδώσουμε και στο θέμα των γλωσσικών γνώσεων. Άρα Πρέπει λοιπόν και να έχουν υψηλό επίπεδο γλωσσικών γνώσεων οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και να μην αποτελέσουν τα υψηλό, οι υψηλότερες προδιαγραφές ε, στη γλώσσα ε, λόγω πρόσβασης, να μην γίνει δηλαδή είτε πιο δαπανηρό, δαπανηρή προσπάθεια να ενταχθούν στο επάγγελμα είτε χρονοβόρα. Επίσης, το θέμα είναι ε, πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάρτιση, αν τα 10 χρόνια ή θα μιλήσουμε για την πλήρη σχολική σταδιοδρομία. Νομίζω ότι ένα καλό σύστημα επαγγελματική κατάρτισης για την υγεία, για τις νοσηλεύτριες, στη Γερμανία ή και την Αυστρία, δεν ε, καλύπτεται με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Γιατί ήδη στη Γερμανία και την Αυστρία έχουμε υψηλότερο επίπεδο κατάρτισης για τις νοσηλεύτριες, με χίλιες ώρες στις φυσικές επιστήμες αλλά και στις επιστήμες του ανθρώπου, στις επιστημονική και άλλες κοινωνικές επιστήμες και ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να ε, αναγνωριστεί ότι έχουν υψηλότερο επίπεδο οι νοσηλεύτριε στη Γερμανία και την Αυστρία σε σχέση, οι νοσηλευτέ στη Γερμανία και την Αυστρία σε σχέση με τι ε, υπόλοιπε χώρε, με 12 χρόνια ουσιαστικά κατάρτιση. Και άρα η παραπομπή στα έτη της κατάρτισης δεν είναι απαραίτητα η σωστή μονάδα υπολογισμού της ε, ισοδυναμίας. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την τροπολογία 460 για το πέμπτο σημείο της περαιτέρω κατάρτισης. Πέραν των κοινών προδιαγραφών για τα επαγγέλματα της υγείας και ιδιαίτερα για νοσηλευτές νοσηλεύτριες, πρέπει να ε, ενισχύσουμε και τις προτάσεις για την περαιτέρω ε, κατάρτιση και προσαρμογή στις επαγγελματικές δεξιότητες. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να το πράξουμε όχι μόνο για λόγους δημογραφικών εξελίξεων και προβλέψεων των δημογραφικών εξελίξεων, αλλά και εν ώψη των εξελίξεων στα επαγγέλματα αυτά και με στόχο βέβαια πάντα την βελτίωση ή την εξασφάλιση της ασφάλειας ε, των ασθενών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο ακόμη μιλητές. Και μετά θα καλέσω την κυρία Βερνιό. Να ολοκληρώσει κυρία Βάιλερ, ευχαριστω πολυ Λίγο ο κύριος Σφάπ. Κυρία ο κυριος Φάπ. Κύριε βαιλερ Πρόεδρε, ευχαριστώ. Φεύγετε, μάλιστα. Καλά. Θα σας πει η κυρία Μίλερ. Λοιπόν, πριν αναφερθώ στο θέμα των νοσηλευτών νοσηλευτριών, θα ήθελα να κάνω δύο μικρές παρατηρήσεις καταρχάς ε, για την κυρία Τσούρονεν και την πρακτική εξάσκηση παρατήρηση που έκανε ήταν ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται εδώ στην, στο τρέχον νομοθέτημα αλλά κάπου αλλού. Μπορώ να καταλάβω τα επιχειρηματά της αλλά από την άλλη η ομάδα των συντονιστών και σκιωδών ε, εισηγητών κάνουν μια προσπάθεια η οποία πρέπει να προχωρήσει, διαφορετικά δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία ενδεχομένω να ρυθμίσουν ε, χωριστά, να δείξουν ενδιαφέρον να ρυθμίσουν χωριστά το ζήτημα της πρακτικής ε, άσκησης, αλλά ε, δεν θα ακολουθήσουν όλα τα κράτη. Αν ακολουθήσουν θα έχουν πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Άρα λοιπόν για την πρακτική εξάσκηση θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο προδιαγραφών, κοινών προδιαγραφών, ώστε να ε, υποχρεώσουμε τα κράτη να αναλάβουν δράση. Για το μηχανισμό επαλήθευσης νομίζω το συζητήσαμε. Απλώς η Επιτροπή ίσως μπορεί να μας εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση τώρα γιατί δεν βλέπω πως είναι δυνατόν να μην έχουμε κανένα μηχανισμό προειδοποίησης σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα. Μπορεί να μας ενημερώσει η Επιτροπή τι είδους ρυθμίσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εάν, παραδείγματι, κάποιο που έχει χάσει την άδεια ασκήσεω συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα κλπ. Τώρα, α περάσω στι ε, νοσηλεύτρε και νοσηλευτέ. Ε, ξέρω ότι η Αυστριακή προχωρούσε τροποποίηση του συστήματός τους και μάλιστα χωρί την Ευρώπη. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε την κοινή αυτή λύση, θα το ρυθμίσουμε μόνο σε Αυστριακή, θα ανεβάσουν από τα 10 στα 12 χρόνια τη διάρκεια των σπουδών. Πιστεύω ότι είναι καλό, καλή προσπάθεια της ηγήτριας μαζί με τους Κιώδης να, να μια συμβαστική λύση. Αλλά για την, στη συζήτηση η κυρία Λεγκρίπ και την ώρα που έμπαινα το είπε, είπε κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ. Παραπέμπει σε μια απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος αλλά αντίστοιχα θα, θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε και στην απόφαση της Επιτροπής Επασχόλησης, πάλι αρμόδιας για γνωμοδότηση. Άρα και τις δύο θα πρέπει ίσως να λάβουμε υπόψη, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι αρμόδια καθήλυνη δική μας επιτροπή, ούτε η ΕΝΒΗ, ούτε η ΕΜΠΛΟ εμείς θα πρέπει να επαληθεύσουμε και να λάβουμε τις αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω ότι μου φαίνεται μάλλον ε, δυσάρεστο να επιλέγουμε να παραπέμπουμε στις θέσεις μόνο της μίας πλευράς. Επίσης ε, είπατε ότι υπάρχουν συστήματα κυρία Λεγκρή που έχουν αποδείξει την αξία τους εδώ και δεκαετίες. Μα και στη Γερμανία έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια πάρα πολλές αλλαγές στις οποίες έχω συμπράξει προσωπικώς, γνωρίζω ακριβώ περί πρόκειται και για το πρόγραμμα σπουδών και για τι αμοιβές αμοιβέ και για το, την οργάνωση του τρόπου εργασία. Άρα μην θεωρούμε ότι στις ε, Βρυξέλ, οι Βρυξέλλε έρχονται να αλλάξουν κάτι το οποίο μέχρι τώρα στη Γερμανία έχει λειτουργήσει χωρί προβλήματα εδώ και 100 χρόνια απαράλλαχτο. Όχι, Μόλι πριν από λίγο καιρό είχαμε μια πρόταση στο αρμόδιο συμβούλιο τη Γερμανία με μια ε, υποχρέωση για μελέτη, για ε, περαιτέρω μελέτη κατάρτιση ε, για όσους ασχολούνται με θέματα υγείας. Ε, μία πρόταση την οποία δεν συμμερίζομαι απαραίτητα, αλλά η οποία έχει ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο και αποδοχή. και από την άλλη πρόταση του Επιτρόπου Μπαρνιέ θα εξωτερώσει αυτό το διπολικό σύστημα της κατάρτισης που γνωρίζει η Γερμανία ε, και το οποίο ενδεχομένω να μην υπάρχει σε άλλα κράτη. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να είμαστε πιο προσεκτικοί στα λόγια μας, να μην φανεί δηλαδή ότι εάν τώρα η Γερμανία υιοθετήσει αυτό που έχουν τα 11 άλλα κράτη σαν σύστημα μπορεί να οδηγηθεί στην καταστροφή. Και επίσης εδώ έρχεται και πρέπει χωριστά να εξετάσουμε τη συζήτηση της διάρκειας των σπουδών 10 ή 12 χρόνια και της κατάρτισης ως, όχι όραμα εν πάση περιπτώσει, αλλά ως στόχο μακροπρόθεσμα. Στη Γερμανία λοιπόν έχουμε όχι μόνο τους εργαζόμενους στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και ε, εκείνους τους νοσηλευτές και νοσηλεύτρες που θα ήθελαν να δοθεί μια νέα όθηση στην Ευρώπη και να αρχίζουν να αλλάζουν κάπως τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ας μην ακούμε μόνο και ας μην παραθέτουμε μόνο τα λόγια της Ένβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε βέβαια να κρίνουμε έτσι τις άλλες επιτροπές, αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ούτως θα περιμένουμε, θα περιμένουμε να δούμε. Ε, μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν τα προσόντα των ανθρώπων και όχι η ίδια η διαδικασία. Ο Σάρβος Βέρπερ ε, θα είναι ο τελευταίος. Ε, μην ε, ξεπεράσετε ε, κοιτάξτε, όσο περισσότερο μιλήσετε, τόσο λιγότερο χρόνο θα έχετε για την επόμενη παρουσίασή σας. Εδώ μιλάμε για τις ε, ε, για τα προσόντα ε, και βεβαίως μακροπρόθεσμα βλέπουμε ότι τελικά παραβιάζουμε τις διαδικασίες κατάρτισης και εκπαίδευσης που έχουν οι διάφορες χώρες. Αλλά βεβαίως... Αυτό βέβαια είναι το όλο πρόβλημα της συζήτησης, όλο αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε σημειώσει, έχουμε ανακαλύψει αρκετές προόδους, αλλά Πρέπει να πούμε ότι έχουν ακόμη πολλέ δυσκολίε να αντιμετωπίζουν ε, οι εργαζόμενοι στον τομέα τη υγεία, νοσηλευτέ, νοσηλεύτε και παρακαλώ να λάβει υπόψη ε, τι ιδιαιτερότητε αυτέ η συγγήτρια. Και για το θέμα των συμβολιογράφων επίση θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να προστατεύει τα συμφέροντα του κλάδου όσο γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. You, you invited, I did say earlier, the Commission is not intervening this time, Barbara, so I'm sure we can get... Μάλιστα, βεβαίω ε, θα έχετε και το χρόνο, θα ακούσουμε τι απαντήσει σα. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Περνατέτ σύντομα για να συνοψίσει όποιε παρατηρήσει ενδεχομένω επιθυμεί. Oui, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριε Βερνιό. Είχα πει ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε τη συζήτηση της νοσηλεύτριας, αλλά βλέπω ότι ε, συστηματικά επανέρχεται το ζήτημα. Είναι βεβαίως σαφές ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολλές εβδομάδες και ενώ προχωράμε πολύ γρήγορα σε άλλα θέματα, πάντα σκοντάφτουμε στις νοσηλεύτριες. Έχουμε διαφωνίες ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων αλλά και ε, με την ε, Κομισιόν. Δεν, δεν θα ήθελα όμως, γιατί αυτό φάνηκε και στη συζητήση με τους σκιώδεις αλλά και σήμερα, δεν, εγώ δεν θέλω ούτε να στιγματίσω της, ε, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, ούτε να στιγματίσω χώρες. Δεν θέλουμε να δείξουμε με, το, με το δάχτυλο ε, χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, άλλες οι οποίες αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες. Δεν το θέλω αυτό. Έχουμε όλοι τον, σαν στόχο την ποιότητα, την ασφάλεια την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτά είναι σημαντικά και πρέπει επίσης να έχουμε όλοι την ε, ε, επιθυμία να καλύψουμε ένα κομμάτι του δρόμου που μας χωρίζει και οι δύο, όλοι, όλες οι πλευρές δηλαδή, και να καθορίσουμε κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας ε, στο καταστατικό της λειτουργίας του, του, του, του επεγγέλματος των νοσηλευτών νοσηλευτριών νομίζω ότι τα κράτη-μέλη, δεν ζητώ, εγώ δεν ζητώ από την Γερμανία να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη το, το εκπαιδευτικό της σύστημα, ε, το οποίο βεβαίως έχει αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερα ποιοτικό. Λέω απλώς για μία ακόμα φορά στους ε, Γερμανούς ότι ε, η Γαλλία, το λέω συχνά ότι η Γαλλία, η χώρα μου, θα μπορούσε ε, να παραδειγματιστεί από την Γερμανία όσον αφορά πολλές εκπαιδευτικές διαδικασίες. Όμως η κινητικότητα των νοσηλευτών είναι μεγάλη. Δεν μπορούμε να το ξεχνούμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ ε, μια κατανόηση από όλους. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε με, με, μεγάλη ε, ταχύτητα, μεγαλύτερη από αυτή που θα μας επέτρεπε ε, να προχωρήσουμε σωστά. Δεν πρέπει να δυναμητήσουμε το μέλλον της Ευρώπης. Οι υπόλοιποι σκιώδεις με την ε, Le Λεγκρίπε, η οποία είναι σκιώδης ε, με το ΕΛΚ, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι παραμένει το ζήτημα των κέντρων αρρωγής που θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Συμμερίζομαι την άποψή της ότι είναι προπαρασκευαστική ε, φάση, δεν συμμετέχει απόλυτα και πλήρως στη διαδικασία αναγνώρισης. Το θέμα των στάζ επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το δούμε και υπό τη σκοπιά της ε, ποιότητας. Όσον αφορά τις επίσημες γλώσσες, ε, νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει ήδη σχεδόν από την πρώτη συνάντηση των σκιωδών ότι δεν πρέπει να ε, πολλαπλασιαστούν οι επίσημες υποχρεωτικές γλώσσες για τα γλωσσικά τεστ. Θα πρέπει να ξαναμετρήσουμε λίγο και τα διακυβεύματα και τις επιπτώσεις γιατί διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο είναι αλήθεια. Το ζήτημα των συμβολιογράφων θα επανέλθουμε γιατί ακόμα το συζητούμε νομίζω ότι θα βρούμε πιο εύκολα ε, συμφωνία για τους ε, συμβολιογράφους. Ο Χριστιανό έφυγε, αλλά ε, πρέπει να, ήθελα να του πω ότι συζητήσαμε, συναντήσαμε συγγνώμη, την μόνιμη ρουμανική αντιπροσωπεία. Συζητήσαμε το θέμα των νοσηλευτών. Όσον αφορά την σιωπηλή ε, ε, άδεια νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει για τις χρονικές προθεσμίες και τα περιθώρια. Ε, για τα στάζ συμφωνώ απολύτως. Τα, τα στάζ είναι η υποχρέωση κατάρτισης στα πλαίσια της κινητικότητας και θα πρέπει να συνδέονται οπωσδήποτε με την επαγγελματική κατάρτιση. Δεν ε, θα κάνει κανείς έτσι ψευτοστάζ, ας πούμε, ή στάζ μαϊμούδες, όπως λέμε στα ελληνικά. Θα πρέπει να είναι ένα στάζ κανονικό, το οποίο θα ε, ε, σχετίζεται με τα επαγγελματικά προσόντα. Όσον αφορά τα γλωσσικά τεστ, Είμαι αναφέρθηκε στο ερώτημα της ε, πρόσβασης ε, στο επάγγελμα πριν ή μετά, πότε πρέπει να γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται αυτά τα γλωσσικά τεστ πριν από την ε, αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός γιατρού, ας πούμε, σε μια νέα χώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φέρουμε ένα γιατρό στην χώρα υποδοχή χωρί εκ των προτέρων να τον έχουμε περάσει από εξετάσει και να ανακαλύψουμε επιτόπου ότι δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα. Όσον αφορά τώρα την επαγγελματική κάρτα, πιστεύω ότι ακόμα και οι δύο δυσκολευόμαστε, γιατί το τα πιλωτικά προγράμματα υπάρχουν, υφίστανται, έχουν αποδείξει, ότι κάτι τέτοιο είναι, είναι ε, ε, θεμητό και μπορεί να γίνει. Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε μελέτες αντικτύπου, οι οποίες και θα επιβραδύνουν τη διαδικασία και θα την κάνουν πάρα πολύ ακριβή, τι να σας πω, ε, αυτό που ε, επιθυμούν οι περισσότεροι εργαζόμενοι του οποίου έχουμε έρθει σε επαφή είναι ότι θέλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουν αυτή τη επαγγελματική κάρτα. Αυτό είναι το, θέμα τους. Ο κύριος ε, Έντζελ τέλο πάντων, λυπούμε δεν θυμάμαι το όνομά σας λέει κυρία Βενιό, είσαστε καινούριο. Euh, euh. Ο κύριος Χέντελ λοιπόν ε, είναι γεγονός ότι φτάσατε τελευταίος, αντικαθιστάτε και κάποιον, οπότε είναι δύσκολα για σας, εν πάση περιπτώσει. Ε, η συνάδελφος έχει δίκιο ότι έγινε ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που με δυσκολεύει λίγο, η έκβαση της ψηφοφορίας δηλαδή ε, με δυσκολεύει, αλλά μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για γνωμοδότηση. Αρμόδια επί της ουσίας και ε, καθήλυν Επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ. Επομένως, ναι, λαμβάνουμε υπόψη την ψηφοφορία της ΕΜΒΗ, αλλά δεν εστιάζω εγώ τη δουλειά μου. Είναι μια ένδειξη για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Από την άλλη πλευρά, εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά. Βεβαίω θα είμαι ε, σε επαφή ε, διαρκώ με την Κομισιόν, την οποία ευχαριστώ που είναι εδώ και που ε, είναι πάντα σε καλή συνεργασία μαζί μα. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο, την Κυπριακή Προεδρία. Όλοι δουλεύουμε με τα ίδια κριτήρια. Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η ποιότητα είναι τα τρία μεγάλα κριτήρια τα οποία συμμεριζόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 23η Ιανουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν λυθεί μέχρι τότε όλα τα θέματα ε, σε λεπτομέρειες, αλλά ελπίζω ότι τα ε, περισσότερα θα έχουν ε, συζητηθεί. Λοιπόν, έχουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για το επόμενο θέμα. Τώρα, εάν θέλετε να φύγετε, παρακαλώ να εγκαταλείψετε την αίθουσα ησύχως. Έχουμε σήμερα κοινή ε, συνάντηση υπό την Προεδρία και ηγεσία του συναδέλφου Σβάμπ. Έχουμε τον κύριο Κιγένσκι. Τα λέω σωστά, σωστά πρόφερα το όνομά σας. Ο κύριος Κιγένσκι είναι εδώ. Um, going to to us. Θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση για την ε, ανάπτυξη ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε σχέση και με την έκθεση του κυρίου Σβάμπ. Έχουμε 120 τροπολογίες ε, που δείχνουν και την σημασία της έκθεσης. Θέλετε να παρουσιάσετε την έκθεσή σας πρώτα ή θέλετε να ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κιλιάνσκι, γιατί έχετε να κάνετε και κάποιε παρατηρήσει όσον αφορά το εξάμεινο. Ε, Σα παρακαλώ να ολοκληρώσετε μέχρι τι 12 το αργότερο. Um, I'm sure it is possible to switch the lights off, yes. No, the slides are coming up. Everything is coming up shortly. Ναι, όλα, όλα τα, όλες τις διαφάνειες θα τις δείτε. Mr. Schwab, just to set the um, I know it's, it, I think it is being booted up for us now. Um, and then we'll ask for... Ωραία. Λοιπόν, μπροστά από τις οθόνες παρακαλώ να μην έχει πολλά φώτα έτσι ώστε να βλέπουμε καλύτερα. And then you can see the slides perfectly in the sunshine. Um, Uh, then I just want to check uh, on the uh, rapporteurs. Mr. is not here. Ο κύριος Κομφεράτη δεν είναι εδώ. Η κυρία Γκέμπχαρτ φαντάζομαι θα μιλήσει εξ ονόματός του. Ευλήν, εσύ εξ ονόματος του και συναδέλφου Κομφεράτη. Πολύ ωραίο ο ο Μάντες δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρούλε είναι εδώ όμως. Και ο κύριος Άφνερ είναι εδώ. Και ο Σέλφος Ντιγιόν είναι εδώ. Έχουμε σκιώδεις, έχουμε ε, ε, άλλους που έχουν πάρει τη θέση των σκιωδών και τους εκπροσωπούν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 Σε 15 λεπτά θα προσπαθήσω να καλύψω την έκθεση για την κατάσταση της ενιαίας αγοράς, την οποία εγκρίναμε χθε ουσιαστικά, δεδομένων των χρονικών περιορισμών. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, ε, να σας δώσω έτσι μια ιδέα για τη δομή ε, και τα βασικά στοιχεία όσον αφορά ε, τους λόγους, ε, θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο έχουμε τόσα πολλά, τόσες πολλές εκθέσεις, έχουμε πολλές εκθέσεις, αλλά σκεφτήκαμε ότι όσον αφορά την ετήσια έρευνα ανάπτυξης και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ε, θα υπήρχε επιτακτική ανάγκη να ασχοληθούμε με τη διάσταση της ενιαίας αγοράς, γιατί όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε όταν βλέπουμε το κεκτημένο και όταν προσπαθούμε να το επιβάλλουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχει επίτηδες ε, δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει στα κράτη-μέλη και να δει που υπάρχουν ε, περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης Γι' αυτό ακριβώς ε, θέλουμε στην διαδικασία της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη να έχουμε μια ειδική ε, θέση για την ενιαία αγορά. Γιατί ο χρόνος ε, των πολλών λόγων έχει παρέλθει, πρέπει να δούμε τι περιορισμούς έχουμε, όλους τους άμεσα επιτεύξιμους στόχους τους έχουμε επιτύχει και προσπαθούμε μία προς μία να εξετάσουμε τις αγορές στα κράτη-μέλη, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα για να δούμε τι προτεραιότητες πρέπει να βάλουμε. Βέβαια αυτό έχει συγχρονιστεί με το κύκλο των ευρωπαϊκών ε, εξαμήνων ε, που τον γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Υπάρχει λοιπόν η δημοσίευση της ε, ετήσιας έρευνας ανάπτυξης, της AGS. Ε, συζητείται στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κάτι το οποίο οδηγεί στα, προγράμματα, στα, στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και μετά υπάρχει ένα δεύτερο κύμα διαβουλεύσεων, οι οποίες ε, σκοπό έχουν τις ειδικέ αναχώρα συστάσεις. Αυτό βέβαια μας φέρνει στη χθεσινή μας, ε, στο χθεσινό κείμενο που εγκρίναμε. Το 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως ε, να ε, κάνει μια παρουσίαση. Θα είναι ετήσια λοιπόν η παρουσίαση που σας κάνω σήμερα. Και στη συνέχεια βεβαίως τον Ιούνιο του 2012 υπήρχε και η ανακοίνωση για την καλύτερη διακυβέρνηση και αναφερόταν η ανάγκη εκπόνησης τέτοιας έκθεσης. Αυτό αυτό είναι το πλαίσιο. Όσον αφορά την ίδια την έκθεση, είναι σύντομη, γιατί ούτω ή άλλως και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ε, πολύ συγκεκριμένα και επί της ουσίας. Ε, δύο βασικά τμήματα υπάρχουν. Το πρώτο είναι μια εισαγωγή, είναι ένα check-up της ολοκλήρωσης. Ε, είδαμε δηλαδή τα δεδομένα ε, στις ε, χώρες μέλη των τεσσάρων ελευθεριών. Μετά εστιάζουμε στη τομείς προτεραιότητας που τουλάχιστον φέτος είναι οι υπηρεσίες, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι ψηφιακές αγορές. Ένα προς ένα, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, προ... Ε, ε, αναγνωρίζουμε τα εμπόδια που υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών. Μερικά παραδείγματα να σας δώσω. Τι εννοώ με την οριζόντια ανάλυση. Ε, προσπαθούμε να δούμε ως προς την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, του κεφαλαίου, των αγαθών ε, και των υπηρεσιών βλέπετε ότι υπάρχει μία πρόοδος που σημειώνεται. Άμα δείτε δεξιά δηλαδή υπάρχει μία πρό, πρόοδος ε, ολοκλήρωση σε σχέση με το 1999. Υπάρχει περισσότερο εμπόριο αγαθών ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε μία τεράστια μείωση το 2009 που είχε να κάνει με την οικονομική κρίση βεβαίως. Υπάρχει πάντως πρόοδος και θα δείτε επίσης στο γράφημα στη δεξιά πλευρά ότι υπάρχει μάλλον ε, μεγαλύτερη ολοκλήρωση με τις ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι εντός, κάτι το οποίο δεν είναι υποχρεωτικά κακό, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι υπάρχει μεγαλύτερο εμπόριο με τις χώρες ε, ε, τις ε, τρίτες χώρες. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες, μπορεί κανείς να το δει με διαφορετικές οπτικές γωνίες, διαφορετικές οπτικές γωνίες Βλέπουμε αναχώρα τι συμβαίνει, βλέπουμε για παράδειγμα πόσες επιχειρήσεις ε, ελέγχονται από μία επιχείρηση σε άλλη χώρα μέλος και βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν διαφορές βέβαια τεράστιες ανάλογα με τη χώρα για την οποία μιλούμε. Στην έκθεση ε, Προσπαθούμε να αναφερθούμε στις διαφορές ε, μεταξύ των κρατών μελών υπ' αυτήν την έννοια. Δεν έχω χρόνο να επιμείνω βέβαια τώρα, αλλά την κάναμε αυτή την, ε, την εστίαση. Σύγκριση τώρα αγαθών και υπηρεσιών. Σε γενικέ γραμμέ θεωρούμε ότι οι υπηρεσίε δεν είναι, υποθέτουμε ότι δεν είναι υπηρεσίες ολοκληρωμένε ε, στο βαθμό που είναι τα αγαθά. Αν δούμε όμως όχι μόνο τα επίπεδα συσχετισμού των τιμών των υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών, αλλά και τις τάσει, ε, ακόμα και στις τάσει υπάρχει έλλειψη συσχετισμού. Οπότε σε κάποια κράτη-μέλη βλέπει κανείς ότι η απόκληση μεταξύ των τιμών των υπηρεσιών σε σχέση με τις υπηρεσίες ε, εκτός της ε, χώρα, αυξάνεται, κάτι το οποίο θα πρέπει να μα ανησυχεί, γιατί ακόμη και αν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μικρότερη ολοκλήρωση αναμένεται μικρότερη ελεκλήρωση στο πλαίσιο των υπηρεσιών από ό,τι στα αγαθά. Ε, τώρα, αυτό που επίση είναι ενδιαφέρον είναι ότι όσο πιο ολοκληρωμένες ε, ε πιο, όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η αγορά στο κράτος μέλος, ε, τόσο φαίνεται αυτό στους καταναλωτές. Δηλαδή έχει, υπάρχει άμεση σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούν ε, οι αγορές των προϊόντων, κάτι το οποίο βέβαια ε, έχει και κάποιες συνέπειες. Αυτά όσον αφορά το εισαγωγικό τμήμα της έκθεσης λοιπόν το check-up, τον έλεγχο της κατάστασης του επίπεδου της ε, ε, ολοκλήρωσης βάσει των τεσσάρων παραδοσιακών ελευθεριών. Μετά περνάμε στους ε, ειδικού τομείς και εκεί επικεντρώνουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει, πρέπει να να αντιμετωπιστούν ως προτεραιότητα. Πρώτα οι, επιχειρή, οι υπηρεσίες, συγγνώμη, γιατί θεωρώ ότι αυτό αφορά περισσότερο αυτή η έκθεση. Βλέπουμε δηλαδή τι προβλήματα υπάρχουν και με την ε, ελευθερία μετακίνησης. Δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες βέβαια. Αλλά για παράδειγμα, αν πάρει κανείς το τελευταίο, τις ε, δοκιμές οικονομικών αναγκών σε κάποια κράτη-μέλη, αν θέλει κανείς να ανοίξει ένα ε, κατάστημα λιανικής πώληση, πρέπει καταρχάς να δει κατά πόσο υπάρχει μια εμπορική ανάγκη για τέτοιου είδους ε, κατάστημα. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν τις βασικές προτεραιότητες, μερικές εκ των οποίων θα είναι η κατάργηση τέτοιου είδους τεστ για την εμπορική ανάγκη για την οικονομική ανάγκη, όπως επίσης και τους περιορισμούς ε, για τα κεφάλαια των επιχειρήσεων κλπ. Θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο ε, στον τουρισμό, στις ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες, στον κατασκευαστικό τομέα, γιατί δείχνουν ότι συμβάλλουν περισσότερο στο ΑΕΠ και έχουν τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο δυναμικό να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη. Να περάσουμε τώρα στον επόμενο τομέα που επιλέξαμε ως ε, τομέα προτεραιότητας. Εδώ έχουμε την ενέργεια και τις μεταφορές. Δεν ε, σας λέω τίποτε το καινούριο, αλλά υπήρχε λίγη μικρή σύγκληση στις ε, λιανικές τιμές, στο αέριο, στον ηλεκτρισμό. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και βεβαίως μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των δικτύων στις μεταφορές. Πάλι μερικά παραδείγματα είναι ε, οι λιμενικές υπηρεσίες κατακαιρματισμένες, ε, ε Υπάρχει επίσης και κατακαιρματισμός του εναέριου χώρου. Προσπαθήσαμε να το, ε, προσπαθούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, το τελευταίο θέμα στο οποίο επικεντρωθήκαμε είναι οι ψηφιακές αγορές. Ε, οι προτεραιότητες εδώ είναι η κάλυψη της ευρείας ζώνης, ειδικότερα ε, σε ε, πιο αραιοκατοικημένες περιοχές, το σύνηθες πρόβλημα του ανεπαρκούς φάσματος και αναφέρομαι κυρίως στην κινητή τηλεφωνία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι και αυτό κάτι το οποίο προωθείται ως ε, μοχλός ε, ανάπτυξης, αλλά υπάρχουν λόγοι και περιορισμοί για τους οποίους ε, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Υπάρχει το πρόβλημα των πληρωμών, αλλά υπάρχει και το θέμα της παράδοσης των προϊόντων, και υπάρχει επίση και το θέμα του αυξανόμενου ανταγωνισμού στι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεδομένων ε, ε, δεδομένου της κρίσεως, επειδή οι ταχυδρομικές υπηρεσίες επενδύουν πολύ περισσότερο ε, στα πακέτα, γιατί αυτό θεωρούν ότι είναι το μέλλον. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές σε επίπεδο ποιότητας και τιμών για την παράδοση των πακέτων, των δεμάτων αν στείλει κανείς κάποιο, κάτι από το Αμβούργο στο Μόναχο ως δέμα, θα σας ε, στοιχήσει πολύ λιγότερο από ότι άμα στείλει κάποιος κάτι από τις Βρυξέλλες στη Λίλη. Δεν έχει σχέση με την απόσταση. Υπάρχει ένα θέμα ε, συνόρων που δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει ένα θέμα ε, που αφορά την ενιαία αφορά, αγορά στον τομέα αυτό. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες, ε, μία ακόμη πρωτοβουλία η υπό την κατηγορία των ψηφιακών αγορών ε, και υπάρχει επίσης και το πρόβλημα της ε, έλλειψης ε, επαγγελματιών στον τομέα της πληροφορικής. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα για τα επόμενά μας βήματα. Εγκρίθηκε χθε ε, η έκθεση, μαζί, ε, το κείμενο αυτό μαζί με την ετήσια έρευνα ανάπτυξη. Είναι μια ετήσια έκθεση, είναι η πρώτη, θα ε, την επαναλάβουμε σίγουρα την επόμενη χρονιά και όπως συμβαίνει συνήθως με τον συνήθη κύκλο της ετήσιας έρευνας ανάπτυξης, θα το συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο, θα το συζητήσουμε στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ε, να ε, φτάσουμε στην αξιολόγηση με τη βοήθεια ε, των κρατών μελών των προγραμμάτων που θα οδηγήσουν στις αναχώρα στάσεις, Τις ειδικές αναχώρα στάσεις. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είχαμε την παρουσίαση αυτή. Ε, και βεβαίως ε, δώσατε και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία χρειάζεται και ο Σάλφος ε, Σφάμπ γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε αυτό το, το θέμα επί του οποίου εργάζεται ο Σάλφος Σφάμπ. Θα ακούσουμε τώρα την έκθεσή σας. Νομίζω ότι έχετε και εσείς κάποιες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε μέσω σχολείων στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη για το 2013. Ευχαριστώ πολύ Μαλκόμ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Είχα αρχικά υπολογίσει να περιορίσω σε τρία σημεία την πρότασή μου, την ε, πρόταση εκθέσεως καταρχάς και τις τροπολογίες. Δεύτερον, την ε, έρευνα, την ετήσια έρευνα ανάπτυξης με την εν λόγω έκθεση που θα έχει σημαντικό ρόλο και τρίτον το ζήτημα των νομοθετικών, ε, της νομοθετικής πρωτοβουλίας, πώς μπορούμε να το καλύψουμε. Μια και έχουμε και λίγο χρόνο. Αλλά θα πρέπει να τοποθετηθώ και στα όσα είπε η Επιτροπή, Πρόεδρε. Αυτό που βλέπω το πολύ θετικό από την παρουσίαση που ακούσαμε τώρα, είναι ότι έχουμε μια πρώτη εικόνα να ενισχύσουμε την διάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς στο ετήσιο, στην έκθεση Αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν χρειαζόμαστε μία παρουσίαση μόνο για το πώς βαίνουν τα πράγματα. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε κάθε φορά, άλλωστε και στο scoreboard, στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. Δεν μας λύνει δηλαδή κανένα πρόβλημα αυτή η έρευνα, η μελέτη. Λίγο πολύ καταγράφει αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Και στη δεύτερη σελίδα ε, βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε καν την προσπάθεια να ενσωματώσει τη δουλειά που είχαμε εμεί κάνει και παρουσιάσαμε πριν από τέσσερι εβδομάδε με τη μελέτη μα για το πώ η δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενό, αφετέρου δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή μα μπορούν να συνδυαστούν. Και μα λέει ότι η ετήσια έκθεση κάνει μια συζήτηση προσανατολισμού κτλ. Αυτό, η συζήτηση προσανατολισμού αφορά το Κοινοβούλιο και από εκεί πέρα δεν εμφανίζεται το Κοινοβούλιο, δεν μα αφορά δηλαδή η έκθεση και γι' αυτό θα έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε διακυβέρνηση της ιστορικής αγοράς εάν παραμείνει η κατάσταση όπως έχει και το λέω για να μιλήσω και για το χρονοδιάγραμμα με το ευρωπαϊκό εξάμεινο που παρουσιάζεται εδώ στην ε, διαφάνεια ότι θα πρέπει στόχος ε, και τη Επιτροπής μας να είναι να ε, μπορούμε τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο το πολύ πολύ με μια πρόταση του, που θα έχει υποβληθεί με τον πίνακα αποτελεσμάτων, το scoreboard δηλαδή για την εσωτερική αγορά, να είμαστε θέσει να ενημερωθούμε για τις εξελίξεις στα επιμέρους κράτη-μέλη, εκεί που είχαν εντοπιστεί προβλήματα προς την υλοποίηση της νομοθεσίας ή με τη, τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, πώς έχει προχωρήσει και έτσι στη συνέχεια με την ε, Annual Growth Survey με την έρευνα της, ε, της έρευνα ανάπτυξης να δούμε τι είδου προτάσει μπορούν να διατυπωθούν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιανουάριο θα ψηφίζουμε σε επίπεδο ολομέλεια στο, ε, πάνω στην πρόταση για τον πίνακα αποτελεσμάτων και θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ε, house specific recommendations, πολύ πιο συγκεκριμένες από αυτές τις οποίες μας παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όπως είπα δεν λειτουργούν, ε, δεν, δεν είναι αποτελεσματικό αυτό το σύστημα, απλώς συνεχίζουμε αυτά που κάναμε το παρελθόν. Γι' αυτό θα ήθελα η έκθεση του Κοινοβουλίου, που έχω εγώ την τιμή να αναλαμβάνω εκ μέρους Επιτροπής μας, να συμβάλλει σε μια συγκεκριμενοποίηση των προτάσεών μας, χωρίς να θέλουμε να θέσουμε κανένα κράτος στο εδόλιο του κατουγερουμένου, να λέμε τι έχουμε αποφασίσει και τι έχει υλοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτέλεσματα. Και πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει, ε, γιατί μόνο αν έχουμε μια ευρή αποδοχή και από την κοινή γνώμη, από τους πολίτες, για τις βέλτιστες πρακτικές και μεθόδους, τότε και αυτό δεν μπορεί να το, στηρίξει σαν προσπάθεια η δική μας η Επιτροπή, τότε μόνο μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει αυτή την προοπτική πιο θετικά. Εγώ είμαι στη θέσή σα. Όλη μα η Επιτροπή ασφαλώ είναι στη διάθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω συζήτηση. Τώρα για την πρόταση εκθέσεω, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. 120 ήταν οι τροπολογίες, το αναφέρατε κι εσείς. Επί της αρχής ε, οι τροπολογίες τουλάχιστον των μεγάλων ομάδων στο σύνολό τους υποστηρίζουν τις κύριες γραμμές της εκθέσεως και αυτό ακριβώς θέλαμε να προσφέρουμε σαν συνεισφορά, δηλαδή η ε, το scoreboard της ενιαίας αγοράς, ο πίνακας αποτελεσμάτων, να καταγράφεται και να αναφέρονται και τα αποτελέσματα, η υλοποίηση, η εφαρμογή, οι ανάγκες για βελτίωση προς την εσωτερική αγορά και σε αυτό να βοηθήσουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο να πείσει τα επιμέρους κράτη-μέλη όπου υπάρχουν δυσκολίες μεταφοράς των οδηγιών, ε, στις προσπάθειές τους, ειδικότερα κράτη τα οποία καθυστερούν ως προς την μεταφορά ή ελείπονται ποιοτικά ως προς την υλοποίηση της νομοθεσίας. Αυτά λοιπόν. Ο κύριος Κοφεράτη δεν είναι εδώ, έχει όμως και εκείνος κάνει προτάσεις. Ε, σε πολλά σημεία συμφωνούμε με τις τροπολογίες, ειδικά στην προσπάθεια να αναπτυχθεί ε, μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς θα προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο πλέον η εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι με τον κύριο Κοφεράτη μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα, δηλαδή μπορούμε να ενσωματώσουμε τις τροπολογίες του στην έκθεση, ώστε να περάσουμε στο Single ε, Market Act υπαριθμών 2, στη δεύτερη νομοθετική πράξη, δηλαδή για την εσωτερική αγορά. Για ορισμένες τροπολογίες χρειάζεται να συζητήσουμε πιο για την υπαριθμό 50 συγκεκριμένα του κ. Κοφεράτη, αν θα πρέπει να παραμείνουμε γενικόλογοι, αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στι προτάσεις μα, αλλά αυτό το συζητάω με τον κύριο Κοφεράτη χωριστά. Επίση, για την κυρία Κέπχαρτη, 107 τροπολογία, η οποία αναφέρεται σε μια ανάλυση εκ των υστέρων post implementation συγκεκριμένα, μετά την υλοποίηση δηλαδή, νομίζω ότι μα βοηθάει ιδιαίτερω και μπορεί να δώσει κάποιε κατευθύνσει για το πώ μπορεί να βελτιώνεται μια τροπολογία. Όταν γίνεται αυτή δηλαδή η ανάλυση μετά την εφαρμογή τη νομοθεσία, μπορούμε να δούμε πιο ξεκάθαρα πού βρίσκονται τελικά οι δυσκολίες επίπεδο κρατών μελών. Το ίδιο και για την 109. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Πρέπει να αναφέρεται η φράση points of single contact για την κυρία Κοράτσα Πίλτ. Ε, πάντοτε αναφέρεται στα retail markets στις, λιανικές, ε, στις αγορές λιανικής πώλησης που βέβαια αποτελούν ένα πολύ καλό δίκτυο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Τώρα αν πρέπει τόσο συγκεκριμένα να τις περιλάβουμε στο κείμενο, ε, ρητά δηλαδή, θα το δούμε. Ίσως πρέπει να το συστήσουμε λίγο περισσότερο. Ο κύριος Διόγκ έχει κάνει κάποιες προτάσεις για διαγραφή. Είναι παρόν εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια σειρά από παρερμηνίε ή παρεξηγήσει για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η έκθεση. Ειδικότερα στην τροπολογία υπαριθμών 1 θα έλεγα ότι... Γιατί βλέπει κανείς την πρόθεση του κυρίου De ότι δηλαδή ο ρόλος της ιστορικής αγοράς μπορεί να είναι και ε, χώρος ανάπτυξης, μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος ανάπτυξης. Αν λοιπόν λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάπτυξη, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την ε, τροπολογία του και γι' αυτό θα συζητήσουμε διμερώς μαζί του. Πάντως θα παρακαλέσω τον κύριο Ντεγιόγκ να μου εξηγήσει στην 37 τροπολογία του ακριβώς τι εννοεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ε, να μην ε, σπέβδουμε, να ε, προξενούμε, να θέτουμε σε κίνηση διαδικασίες προσβολής επί παραβάση των συνθήκων. Από την άλλη δεν μπορούμε και να επαναπαυόμεθα και να μην αναλαμβάνουμε καμία δράση, να αποκλείουμε εκ προημίου την ανάληψη κάποιας δράσης δικαστικής. Πάντως ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειες και προσβλέπω σε καλή συνεργασία για την έκθεση και για την ετήσια έκθεση ανάπτυξης που μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει μια έκθεση ολοκλήρωσης η οποία στηρίζεται στι βασικέ ελευθερίε, προσανατολίζεται καταρχά στι βασικέ ελευθερίε, βασικέ ελευθερίε, αλλά ε, αναφέρεται και σε κάποια επιμέρου θέματα, όχι τα ίδια κάθε χρόνο. Μα δίνει πληροφορίε, οι οποίε είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Επί παραδείγματι, στι καθυστερήσει ε, πληρωμών πάντα οι ίδιε δημόσιε υπηρεσίε, οι αρχέ είναι οι ίδιε ε, που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πληρωμών, εξοφλήσεων των υποχρεώσεων του. Άρα νομίζω ότι έτσι μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα, μπορούμε να διαπιστώσουμε πού εγγύνται τα προβλήματα, πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τη στηρίξουμε στην προσπάθειά της αυτή. Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να είναι πιο συγκεκριμένη στα παραδείγματα που προσφέρει και σε παραδείγματα που ενδεχομένως έχει να, να δώσει και προτάσεις πάντως, εμείς θα λάβουμε τις εκθέσεις ανακράτος country specific ε, τον Ιούνιο και τις σχετικές συστάσεις εμείς θα τις διατυπώσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο της οδηγίας έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε πώς προχωρεί η διαδικασία ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο σε επίπεδο κρατών μελών. Και Πρόεδρε, κλείνοντα, θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ στην έκθεση με κάποιε τοποθετήσει επί τη αρχή. Έχουμε λοιπόν ε, μέχρι τι 6 ε, Δεκεμβρίου την προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών. Ε, θα πρέπει ωστόσο να έχουμε τη δυνατότητα χάρη τροπολογίε αυτέ να πούμε πέντε λόγια για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη, για την έκθεση ολοκλήρωση και έτσι πρέπει να μα δοθεί δυνατότητα να καταθέσουμε επιπλέον τροπολογίε. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα συμπεριλάβουμε τα πάντα μέσα. με την επιπλέον δυνατότητα λόγω των προθεσμιών θα πρέπει μόνο στα αγγλικά να είναι δυστυχώ τροπολογίε, αν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν να καταθέσουμε μια έκθεση νομοθετική πρωτοβουλία, ιδέα πρωτοβουλία, ως ε, κοινοβούλιο. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ξέρω ότι οι υπηρεσίες μας, η γραμματεία έχει ξεπεράσει κάθε τεχνικό εμπόδιο ως προς το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω εάν η Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να λάβει υπόψη μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, εν προκειμένου προβλέπεται α, η δυνατότητα από τις συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσει για κατευθυντήριες γραμμέ ε, προ το Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα, τα προτελευταία χρόνια. Εάν λοιπόν πρόκειται να κατατεθούν τροπολο... ε, γραμμές και το Κοινοβούλιο μόνο γνωμοδότηση μπορεί να διατυπώσει, τότε ε, πάλι δεν έχει αξιοποιήσει αυτή νομική βάση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά μπορούμε την ε, νομική αυτή βάση να την αξιοποιήσουμε εμείς για έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας. Και έτσι με το άρθρο 14 και ε, σχετικά με τις συστάσεις της επιμέρους για τα κράτη μπορούμε εμείς να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για νομοθετική έκθεση ως κοινοβούλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ίσως μπορέσουμε να βοηθήσουμε για καλύτερη διακυβέρνηση στην εσωτερική αγορά, να συμβάλλει το κοινοβούλιο με τις δικές του ιδέες. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευρύτατη αυτή παρουσίαση του πώς θα συνεχίσουμε, γιατί ε, πρέπει όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με την ουσία της έκθεσης και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνάδελφοι δείχνουν τόσο ενδιαφέρον. Λίγο ακόμα σχόλια και μετά να μιλήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Κυρία Γκέπχαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Σφάπ, Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου κ. Κοφεράτη, ο οποίο είχε μια πολύ σημαντική δέσμευση στην ε, Ιταλία και δεν μπόρεσε να έρθει. Εχθέ με εκπροσώπησε εκείνο γιατί είχα εγώ αντίστοιχη δέσμευση στην ε, Γερμανία. Ε, πότε πότε συμβαίνουν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμω, που θα τον εκπροσωπήσω εγώ σήμερα. Ο κύριος Κοφεράτη λοιπόν με παρακάλεσε να επισημάνω μια σειρά από ζητήματα, αλλά πρώτα θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια ως προς την ετήσια έκθεση ανάπτυξη του 2012 που παρουσιάστηκε νωρίτερα και θα ήθελα να πω τα σχόλιά μου είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη δική σας, με σας κύριε Σφάπ. Πρέπει να πω ότι με απογοήτευσε παρουσίαση που λάβαμε. Λίγο πολύ τα ίδια πράγματα με αυτά που είχαμε ακούσει και πέρσι μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα καινούριο μέσα σε ένα χρόνο, τι θα περιμένουμε για τον χρόνο; για τον επόμενο χρόνο, αν έχουμε πάλι την ίδια προσέγγιση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια προσπάθεια παραπάνω. Για δε την ε, εκτίμηση ότι περιμένουμε κάτι διαφορετικό στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξέφρασε ο κύριος Σφάπ, θα τη συμμεριστώ και εγώ. Και εδώ θα επαναλάβω μια πολύ ωραία φράση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μου άρεσε, αλλά που πιστεύω θα πρέπει και να γίνει πραγματικότητα, να μείνει στα λόγια μόνο. Αυτό που είπε δηλαδή ότι τέλειωσε η εποχή των μεγάλων ε, λόγων και ότι πια πρέπει να περάσουμε στα έργα. Μακάρι, μακάρι να το δούμε και στην πράξη αυτό. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και υλοποίηση. Και θα ήθελα να σχολιάσω με ένα, μία φράση που με παραξένεψε πρέπει να πω το θέμα των ταχυδρομείων και τις διαφορές στο τιμολόγιο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό οφείλεται απλώς και μόνο στην απελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ή τα ταχυδρομεία είναι ε, ελεύθερα να αποφασίσουν τι είδου τιμολόγιο θα επιβάλλουν για κάθε διαδρομή. Θυμάμαι πολύ καλά τις διαφωνίε όταν είχαμε ισότιμα τιμολόγια μεταξύ και Γερμανίας, αλλά μετά την απελευθέρωση έγινε αλαλούμ όλο το θέμα των ε, τιμολογίων. Συνέπειε αυτών που αποφασίστηκαν πριν από κάποια χρόνια είναι οι διαφορετικές τιμές. Όταν είναι λοιπόν οι τιμές ίδιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισότιμες, τότε ίσως θα ήταν καλό να μην προχωρούμε σε απελευθέρωση πάση θυσία, για να διατηρούμε αυτές τις καλές τιμές. Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει όμω, μάλλον δεν είναι ρεαλιστικό το να ζητούμε κάτι τέτοιο. Το μέχρι εκεί φτάνω ακόμα κι εγώ να το αναγνωρίσω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μια άλλη διαπίστωση αντίφαση στην ε, αξιολόγηση υπηρεσιών, των αγορών των υπηρεσιών. Σελίδα 10 στην παρουσία σας, όπου μας λέτε ότι οι διπλές ρυθμίσεις και οι αβεβαιότητες ε, σχετικές με τους ε, κανόνες, την εφαρμογή των υπηρεσιών κτλ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Αλλά ταυτόχρονα εσείς, μάλλον το δίκαιο το ευρωπαϊκό έχει προσφέρει τη δυνατότητα για ένα επικουρικό σύστημα ή ένα ε, εκούσια συμμετοχή σύστημα. Επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί σας ενοχλεί εφόσον αυτό έχετε προβλέψει εσείς. Γιατί το καταδικάζετε λοιπόν, γιατί το λέτε ότι δεν είναι καλό. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς αυτό έχετε προβλέψει, προτείνει, υλοποίηση. Ξέρω ότι πολλά πράγματα έχουμε να συζητήσουμε και περιμένω να γίνουν αυτές οι συζητήσεις με τους συναδέλφους. Κατά τα άλλα, ε, συμφωνώ με τον κύριο Σφάβο και με τον κύριο Κοφεράτη ε, ότι πρέπει η εσωτερική αγορά, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αποτελέσει ένα κεντρικό σημείο, τον πυρήνα ίσως του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί. Όπως πρέπει να ενισχυθεί και η πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως εν ώψη της ε, κρίσης που αντιμετωπίζουμε τώρα στην οικονομία, στις εθνικές οικονομίες. Και επίση, όπω ε, πρέπει να πω, είναι πολύ σημαντικό για εμά του σοσιαλδημοκράτε και τον κύριο Κοφεράτη, ιδιαίτερα τον ενδιαφέρει. Το βλέπουμε άλλωστε και από τι τροπολογίε που έχει καταθέσει στην, πρόταση σας, στην έκθεση σα, κύριε Σφαπ. ότι δεν ε, αρκεί μόνο το να δίνουμε έμφαση στην προστασία των καταναλωτών και των επιχειρηματιών, όπου συμφωνούμε απολύτως μαζί σας, αλλά πρέπει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να υπογραμμιστεί η σημασία της προστασίας του πολίτη και του εργαζομένου. Πρέπει και αυτό να το βάλουμε μέσα στο κείμενο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριο Κοφεράτη επίση, ε, στι ε, σημειώσει που μου έστειλε, τι οποίε δεν θα σα αναγνώσω γιατί διαφορετικά θα μου είναι πολύ ώρα, αλλά θα επισημάνω ορισμένα σημεία. Μου λέει λοιπόν ότι συμφωνεί με την ιδέα της ε, νομοθετικής πρότασης με βάση το 23 του 114 της συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμά, τους δημοκράτε είναι η σωστή λύση και επίσης η ενσωμάτωση της εσωτερική αγοράς στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και να το ξαναπώ και κυρίως με προοπτική την Ευρώπη του 2020 πρέπει να είναι ενισχυμένη. Συμφωνεί λοιπόν με την υπογράμμιση αξίας εσωτερικής αγοράς με τους πέντε τομείς που θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα και πάλι, όπως είπα, η προστασία του καταναλωτή, του εργαζομένου, τα δικαιώματα του πολίτη. Για το ε, Single Market Act υπαριθμών 2, το δεύτερο νομοθέτημα για την εσωτερική αγορά, με καλύψατε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα ίδια. Ο κύριος Σκοφεράτη νομίζω είναι διατεθειμένος και έτοιμος για πολύ καλή συνεργασία μαζί σας και στο μέλλον και βεβαίως να προσφέρει χείρα βοηθεία στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για να βελτιώσει τη δική έκθεση. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει τη δική της έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την έκθεση. αν πρόκειται να γίνει μία ε, ετήσια έκθεση, τότε πρέπει να έχουμε και εμείς να τη συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των εκθέσεων. υπάρχουν ζητήματα για το πώς θα συνεχίσουμε και πώς ε, θα δράσουμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ουσία του πράγματος και ε, να ξέρουμε τι θέματα θα πρέπει να επιλύσουμε. Έχουμε 10 λεπτά για να ακούσουμε για τους κοιόδης συζητητές. Συγγνώμη, δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα. Έχουμε τέσσερις σκιώδεις εισηγητές ε, και έχουμε και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε. Δύο λεπτά ο καθένα έχετε. Θέλω να δώσω και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν είναι όμω ο μοναδικό γύρο συζητήσεων. Θα μπορούσα να είμαι σύντομο, ε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την έκθεση του Αντρέα. Του ή άλλω είναι μια, συζη... μια γραμμή που την έχουμε συζητήσει εδώ και χρόνια. Είναι καλό να έχουμε νομοθεσία επί του θέματο αυτού. Κρίμα που δεν είναι εδώ. Ε, η Κρίστεν, γιατί θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο θέλει να ε, διαγράψουμε την ε, έννοια του κανονισμού. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ε, συζητήσει, αλλά εξακολουθώ να έχω την απορία. Θα τη ρωτήσω την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέτειο της εγκαθίδρυσης της ενιαίας αγοράς, όμως δεν υπάρχει συνεργασία γιατί μόνο όσοι βρίσκονται εδώ ε, ξέρουν ότι είχαμε την επέτειο και οι κουρτίνες ήταν κλειστές εν ολίγης, ε, είναι σαν να ντρεπόμαστε, σαν να φοβόμαστε να πούμε στον κόσμο εκτός του κτηρίου ότι δουλεύουμε ε, για εκείνους. Ε, εμείς θα θέλαμε και στην Ολλανδία να οργανώσουμε μια εκδήλωση για την επέτειο αυτή 90 άτομα μέσα στη συνεδρίαση το ήξεραν, μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης, αλλά εκτός δεν το ήξερε κανείς εγώ παραπονιόμουν ε, ε, για, την, ε, για, το γραφείο πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για να μπει κανείς πρέπει να έχει badge, διαφορετικά δεν μπορεί να μπει. Αν θέλουν όμως να είναι πιο ανοιχτοί στο κοινό, πρέπει να είναι ανοιχτά τα παράθυρά τους, ανοιχτή η πόρτα τους, για να δείχνουν στον κόσμο πώς δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι δουλεύει για τον κόσμο. Όχι να είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να μπει κανείς. Είμαστε τόσο ε, απασχολημένοι και απορροφημένοι από τη δουλειά μας, δεν επικοινωνούμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα αρχίζουμε δηλαδή ε, να βλέπουμε ε, τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ίσως θα έπρεπε να δουλέψουμε μαζί με τη Ρόζα γιατί αυτό που κάνανε στην Πολωνία ήταν ότι πήγαν εκείνοι στον κόσμο και δεν κάλεσαν τον κόσμο να έρθει στις Βρυξέλλες που είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Αλλά τέλος πάντων κάτι άλλο ήθελα να πω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα αυτά που άκουσα από τον κύριο Σφαμπ. Έτσι που μας τα είπε δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Πάντα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει μεγάλα άλματα δεν πάει τα πράγματα μέχρι εκεί που πρέπει να πάνε. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ορισμένα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια έκθεση πρωτοβουλία. Συμφωνώ απολύτως με αυτήν ε, την ε, πρόταση. Κυρία Μακλάρκεν, ε, η ενιαία αγορά είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι η εφαρμογή της, η πραγματική εφαρμογή της έχει άμεσα αποτελέσματα στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Εμείς συμφωνούμε με την νομοθετική προσέγγιση και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σφαμπ για την έκθεσή του. Κάποιες τροπολογίες πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν και γι' αυτό τις υπέβαλα. Όσον αφορά το τεστ ε, της ε, ενιαίας αγοράς, ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε με καλύτερο τρόπο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας νομοθετικής πρότασης για τη λειτουργία της ε, ενιαία αγοράς. Δεύτερον, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο δημοσίων υπαλλήλων ε, στα κράτη-μέλη για να τους βοηθήσουν ε, να εφαρμόζουν καλύτερα την ενιαία αγορά. Μιλάω πέρα από το Solvit. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχω και εκεί κάποιε παρατηρήσει, αλλά μπορούμε να τι συζητήσουμε αργότερα. Συμφωνώ όμω απολύτω και σα υποστηρίζω πλήρω την προσέγγιση σα, κύριε Σφαμπ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα μπορούσα να είμαι σύντομο. Η δική μας άποψη είναι κατά τη διαφορετική. Για το στόχο συμφωνούμε. απολύτω πλήρης μεταγραφή των διατάξεων της ενιαίας αγοράς ε, και για μας αυτό αποτελεί στόχο. Υποστηρίζουμε τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν όμως δει κανείς το οικονομικό εξάμεινο, ένα από τα σημαντικά προβλήματα που έχει η ομάδα μας με το οικονομικό εξάμεινο είναι η έλλειψη εστίασης ε, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο του εξαμεινού Αυτό που κάνουμε είναι ότι τονίζουμε την ενιαία αγορά, δεν έχουμε ένα παρόμοιο σύστημα για τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις υποχρεώσει. Ε, δεν έχουμε διασφάλιση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς για τα κοινωνικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια ρήτρα κοινωνική πρόοδου. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι κάπως ε, παράτερο να επικεντρωνόμαστε σε ε, μία πτυχή και να μην αναφερόμαστε στις υπόλοιπες πτυχές ε, τις οποίες μόλις ανέφερα. Για τη γρήγορη διαδικασία, για τις διαδικασίες επί νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε κάτι τέτοιο και για την εσωτερική αγορά, αλλά ε, θα έπρεπε να ισχύει και για τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, αν δει κανείς τις προκλήσεις της κλιματικής ε, αλλαγής ε, ενώπιών μας. Υπάρχει και εκεί μια ανάγκη ε, επίγουσα. Δηλαδή να ρυθμίζουμε κάτι σε ένα σημείο όταν θα, μπορούσε να θα έπρεπε να είναι οριζόντιο, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Συμφωνώ σε γενικέ γραμμέ με την προσέγγιση του κύριου Σφάντα, αλλά έχω πολλέ ανησυχίε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ε, πρώτη. Άννα Μαρία, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ, να ευχαριστήσω και να επικροτήσω την έκθεση του κυρίου Σφαμπ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τρεις λόγους. Πρώτον, ε, το συνδέει περισσότερο με την, ε, το πρόγραμμα ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση ένα μήνυμα προ τα κράτη-μέλη ότι φτάνει πια. Νησάφι. Ότι πρέπει να περάσουμε στη δράση. Όταν λέμε ότι ε, κάνουμε απλώς μία δήλωση ότι τι ωραία που είναι η ενιαία αγορά, οι υπηρεσίες είναι πάνω από 65% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε 2,6% επιπλέον να ε, κερδίσουμε ε, τα προηγούμενα πέντε χρόνια αν ε, ήταν σωστή εφαρμογή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στα κρατημέλη ότι η μεταγραφή, η επιβολή και η εφαρμογή της ενιαίας αγοράς είναι πραγματικά κρίσιμη και ελπίζω να ε, υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου προς την κατεύθυνση της μηδενικής ανοχής για τη μη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Ναι. Θα το έλεγα και εγώ αυτό. Έχει άμεση σχέση με τη δική σας έκθεση που προηγουμένως χθες τη συζητήσαμε. Βέβαια, καταλαβαίνουμε την ε, μεγάλη σημασία των υπηρεσιών που αναφέρονται πάρα πολύ στις εκθέσεις σας. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να πάρετε το λόγο κυριαρίας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρώ είναι εξαιρετική η δουλειά σας. Πρέπει να διαγνώσουμε πρώτα τα προβλήματα πριν προτείνουμε λύσεις και συγκεκριμένες δράσεις. Αυτό όμως με απασχολεί είναι ένα πράγμα συγκεκριμένο. Στη σελίδα 14 μιλάμε για ψηφιακές αγορές στον πληθυντικό. Πάντοτε όμως λέμε λέγαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε μία ενιαία ψηφιακή αγορά. Δεν συμφωνούμε λοιπόν με την πληθώρα ψηφιακών αγορών. Μία είναι η ψηφιακή αγορά. Μάλιστα λέει ο πρόεδρος. Η έκθεση και η παρουσίαση της ε, έθεσε πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σήμερα. Άρα πρέπει να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σφάμπ ε, και θα πρέπει να δώσω ξανά και το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απλώ θα ήθελα να πω και εγώ κάτι πολύ σύντομο. Ένα από τα απογοητευτικά πράγματα στην έκθεσή σα και έχει άμεση σχέση με αυτό που υπόθηκε για το γεγονό ότι είμαστε πολύ εσωστρεφεί και ομφαλοσκοπούμε τέλο πάντων ελαφρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν έχουμε τίποτε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, ε, ούτε από τη Μεταφορών. Α, έχουμε κάτι από την Επιτροπή Μεταφορών. Α, πάλι καλά. Κάτι είναι και αυτό. Τουλάχιστον η Επιτροπή Μεταφορών ε, κινητοποιήθηκε. Έχουμε κάποιες ε, τροπολογίες πράγματι. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Το θέμα της ανεργίας επίσης. Ε, υπάρχει ένα ξεχωριστό τμήμα απασχόλησης ε, που αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να ασχοληθούμε με αυτό. Οι συντονιστές μου το ε, είπαν ξεκάθαρα αυτό. Ο κύριος Φαμπ. Ναι, πολύ σύντομα πρόεδρε, δύο σημεία. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω του συναδέλφου για όλε τι παρατηρήσει, τι επισημάνσει και να καταστήσω σαφέ ότι για μένα η εσωτερική αγορά είναι πολύ περισσότερα από ότι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά. Όσον αφορά λοιπόν τη διακυβέρνηση τη εσωτερική αγορά, βεβαίω και μπορούμε να συζητούμε. Πιστεύω όμω ότι εάν επικεντρωθούμε στην εσωτερική αγορά, τα κοινωνικά στοιχεία, τα περιβαλλοντικά στοιχεία θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίση. Εάν λοιπόν η, οδηγία για τις υπηρεσίες μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές για τους ε, ε, πολίτες, για τους καταναλωτές, προφανώς αυτό έχει και κοινωνικές συνέπειες. Εάν δεν υλοποιείται σωστά η οδηγία αυτή, και δεν είναι καλές οι τιμές, πάλι, δεν, πάλι έχει κοινωνικές συνέπειες. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα μπορούσαμε να σωματώσουμε σε μια συζήτηση για την εσωτερική αγορά, αλλά κάπου πρέπει να θέσουμε και κάποια όρια. Εδώ μιλούμε λοιπόν για την νομοθεσία της σχετική με την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και ως εκ τούτου για θέματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά και άλλα. Ε, επίσης ε, μέχρι 6 Δεκεμβρίου, όπως είπα, έχουμε τη δεύτερη αυτή προθεσμία για τροπολογίες. Ε, μέσα σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για να δούμε το θέμα του, της μορφής ε, νομικά, αν θα πρόκειται για έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να λάβει κάποια πρωτοβουλία και μέσα στα Χριστούγεννα θα έχουμε το περιθώριο να ξανασκεφτούμε όλα αυτά και να δούμε τι άλλο μπορούμε να προσφέρουμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ευχαριστώ πολύ. Um, Σας ευχαριστούμε πολύ. θα έχουμε ε, συμβολές υπομορφήν ε, τροπολογιών για το στοιχείο της εσωτερικής αγοράς που αναφέραμε όλοι προηγουμένως. 6 Δεκεμβρίου να έχουμε τις τροπολογίες αυτές. Ελπίζω ότι οι συντονιστές θα θέλουν και αυτοί ε, ως εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων να ενισχύσουν την κατάσταση και θα συζητήσουμε και με τον κύριο Μπαρνιέ βεβαίως ο οποίος θα έρθει ή θα κάνουμε μια, θα στην Επιτροπή, θα έχουμε μια χωριστή ε, συνάντηση μαζί του, θα δούμε. Ευχαριστώ ε, όλους. Κλείνουμε ε, και την συνεδρίαση δεν ε, ε, γίνεται πλέον, ε, δεν μεταδίδεται πλέον. Έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας τον Δεκέμβρη, αλλά πριν να σας πω ότι έχουμε μια εσωτερική συνεδρίαση σήμερα το απογεύμα, έτσι ώστε να μιλήσουμε και για, την... για όλα τα μελλοντικά μας ζητήματα. Ευχαριστώ.